στις 12. Επόμενο θέμα είναι η έκθεση Ντελάνγκε για την επισητιστική κρίση. Έχει το λόγο η κυρία Ντελάνγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενώ οι περισσότεροι συνάδελφοι προφανώς και τρώνε βραδινό αυτή τη στιγμή, θα ήθελα ωστόσο να θίξω ένα πολύ σημαντικό για τη γνώμη μου ζήτημα, επί το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ασκαιώτες συζητητέ από τις άλλες πολιτικές ομάδες για την πολύ καλή συνεργασία. Ε, με στήριξαν κατά τη συγγραφή αυτή τη ε, ε, έκθεση και μάλιστα ψηφίστηκε ομόφωνα στην Επιτροπή στην Αρμόδια ε, Είχαμε πρόσφατα πολλά σκάνδαλα, μεταξύ του οποίου και το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τέτοιο ζήτημα. Ε, πρώτο στοιχείο που εντοπίζουμε είναι η έλλειψη ε, αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων. Βάσει των ελάχιστων διαθέσιμων μελετών, και από τα στοιχεία της Europol γνωρίζουμε τουλάχιστον ε, περί τίνος πρόκειται. Γιατί ε, προϊόντα για το κρέας, το ελαιόλαδο, ακόμα και το, ο καφές στο τσάι. Ξέρουμε ότι αυτό το σκάνδαλο, αυτά τα σκάνδαλα ε, πλήττουν εκατομμύρια πολίτες και επιτέλους και οι αρχές αρχίζουν να ενδιαφέρονται. Όμως υπάρχει σημαντική αναγκαιότητα να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Αυτή είναι η πρώτη μας απέτηση. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει έναν ενιαίο ορισμό της απάτης στα γεωργικά τρόφιμα και κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει. Η έκθεση αυτή είναι το πρώτο βήμα. Βρισκόμαστε λοιπόν στα πολύ πρώιμα στάδια αυτής της διαδικασία. Και πολλές φορές ε, δεν ε, επενέβησαν επαρκώς οι ευρωπαϊκές αρχές, ιδίως εκεί όπου δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος, ε, άμεση απειλή για τη δημοσία υγεία. Όμως ε, ε, αυτό πλήττει πέραν των καταναλωτών, κλονίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει και όλους τους υπόλοιπους φορείς και εργαζομένους που απασχολούνται στον τομέα. Ο κίνδυνος της ε, απάτης ε, στα γελικά τρόφιμα καθορίζεται και από το ενδεχόμενο κέρδος και από τον κίνδυνο να τον πιάσουν κάποιο στα βράσα. Για παράδειγμα, το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου στην Ιρλανδία. Τέσσερις επιχειρήσεις συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Τρεις επιχειρήσεις ξεκίνησαν ε, ακριβώς έξω από την Ιρλανδική επικράτεια. Έμεινε μόνο μία επιχείρηση που ε, μπορούμε λοιπόν, ε, ε, εναντίον της οποίας μπορούμε να κινήσουμε δίωξη. Και η δίωξη αυτή θα αφορά ουσιαστικά μόνο 30.000 ευρώ ενώ το κέρδος είναι 65.000 ευρώ μόνο για ένα κοντέινερ που περιέχει κρέας αλόγου αντί για βόλιο. Πρέπει πολλά λοιπόν να αλλάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, πιο αυστηρέ ποινέ. το διπλάσιο της, του ενδυνάμει κέρδου και για όσους ε, διαπράττουν το ίδιο αδίκημα πολλές φορές θα πρέπει να τους αφαιρείται η άδεια. οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να έχουν μια καλύτερη προσέγγιση, να είναι λιγότερο προβλέψιμη προσέγγιση τους, περισσότερο ε, να ακολουθεί το παράδειγμα των αστυνομικών αρχών όπως συμβαίνει και στη Δανία και στην Ιταλία. Καλύτερη συνεργασία με την Europol, με το νέο σύστημα ειδοποιήσεων. Με ένα τέτοιο παζλ 28 κρατών μελών για να διαμορφώσουμε μία ενιαία εικόνα είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχουμε καλύτερες, καλύτερα στοιχεία ε, και σε ό,τι αφορά τους εμπόρους και το καθεξής, αλλά και ε, τι υπεραγορέ. Το να λέμε κάθε φορά ότι χρειαζόμαστε πιο φτηνά προϊόντα δεν επιφέρει και καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα. Η έκθεση πολύ σωστά αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά την επισήμανση θα μπορούσε, λένε κάποιοι, να, να υπάρχει απάτη παρά την επισήμανση. Όμως, καλύτερο είναι να έχουμε επισήμανση για να γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα που αγοράζουμε, ιδίως αγοραζουμε ιδιω πρόκειται για κρέας. Έτσι έχουμε και μια αξιολόγηση αντικτύπου και ε, αποφεύγουμε και το περαιτέρω διοικητικό άκθος. Επομένω, περιμένουμε την ε, αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστούμε κυρία Αντελάγκε. Διαδικασία Κάτσδιάη. Πρώτος μιλητής, ο κύριος Σέιερ. Η κυρία Σέιερ. Το... Το ψήσιμο αυτό ξεκίνησε από το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου και Επιτροπή σωστά συζήτησε το θέμα των διαθροτικών προβλημάτων στην αγορά τροφίμων. Αυτή τη στιγμή η επισητιστική κρίση είναι ε, σοβαρή, διότι η εμπιστοσύνη στην αλυσίδα διατροφής έχει αποδυναμωθεί σοβαρά. Εμείς πουλάμε τρόφιμα με εικόνες καθαρότητας. Ωστόσο, παρότι μάλλον η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα της επισήμανσης, τούτο δεν οδηγεί σε σωστούς ελέγχους και σε εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Ο έλεγχος λοιπόν θα πρέπει να εξετάζει πάντα τους κινδύνους απάτης. Ο κύριος Πίκουλα. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την έκθεση σχετικά με την επιστημιστική κρίση, την απάτηση στην αλυσίδα των φήμων και τη διενέργεια ελέγχων. Θέλω να τονίσω ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα από το σκάνδαλο κρέατος αλόγου Υποστηρίζουμε λοιπόν την καταπολέμηση της απάτης στην αλυσίδα τροφίμων. Έχουμε σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η Κροατία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους ε, στην εισαγωγή κρέατος. Σήμερα έχουμε ανοίξει την αγορά μας ε, στις εισαγωγές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπιστοσύνη ωστόσο των κρατών ε, καταναλωτών κινδυνεύει να χαθεί εάν διαπιστωθεί απάτη. Εμείς υποστηρίζουμε αυστηρότερους ε, ελέγχους και εντατικότερη καταπολέμηση της απάτης στο σημαντικό αυτό κλάδο. prevare u prehrambenom lancu problem s kojim se moramo oštro Η απάτη στην ε, διατροφική αλυσίδα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ αυστηρά γιατί οδηγεί στην ε, μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στην, ε, σε βλάβες, σοβαρές βλάβες της δημόσιας υγείας. Επίσης, Ε, ε, τα φαινόμενα απάτης ε, στα τρόφιμα έχουν πολλαπλασιαστεί και οι επιθεωρήσεις είναι ανεπαρκείς. Πολλά προβλήματα υπάρχουν στην αλυσίδα διανομής και πολύ συχνά έχουμε προϊόντα χαμηλής ποιότητας, τα οποία είναι πιο ανταγωνιστικά και ε, όσο θα πρέπει να φροντίσουμε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έχουν σημειωθεί πάρα πολλά σκάνδαλα σε αυτό το χώρο. Στη δική μου χώρα είχαμε το σκάνδαλο με το κρέας ε, αλόγου και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό θα πρέπει να πούμε ότι η εγρήγορση των αρχών οδήγησε στην διαλεύκανση του σκανδάλου ε, και οδήγησαν ε, στον περιορισμό αυτού του φαινομένου που ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Ντελάγκ ανφέρθηκε ένα πολύ σημαντικό σημείο όταν αναφέρθηκε στις κυρώσεις. Όποιες κυρώσεις και αν ε, επιβάλλονται αυτή τη στιγμή θα πρέπει μελλοντικά να διπλασιαστούν ή να τριπλασιαστούν. Ε, αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του φαινομένου. Η επαγρύπνηση είναι βεβαίως ιδιαίτερο σημαντική καθώς και το ζήτημα της ορθής σήμανσης και της ε, ορθής ε, ιχνηλάτησης ε, των προϊόντων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερως για το κρέας αλόγου αλλά και για τα άλλα είδη τόσο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σα πω ότι έχω σταματήσει να τρώω κρέα εδώ και δύο χρόνια, οπότε αυτά τα θέματα με αφορούν ελάχιστα. Κυρία Σεναλόβο účinně řešit opakující se αυτή τη κρίση με το αλογίσιο κρέα, Ίσως να λυθεί αυτό το διαρκές πρόβλημα της απάτης στα τρόφιμα και η υπεραπίση των ετικετών στον τομέα των τροφίμων. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς από πού προέρχονται τα εν λόγω προϊόντα και όσοι χρησιμοποιούν παραποιημένες ετικέτες, ψευδείς ετικέτες, ε, πρέπει να υποστούν κυρώσεις. Επίσης υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συσκευασία είναι μία πτυχή, αλλά το περιεχόμενο είναι μία δεύτερη πτυχή. Κάτι θα ήθελα να ε, ζητήσω. Οι προτάσεις και τα παράπονα των καταναλωτών πρέπει να διερευνώνται διότι ακούμε διαρκώς τη ίδια παράπονα. Η ποιότητα είναι και ένα θέμα προτίμησης, είναι κάπως υποκειμενικό ζήτημα. Δυστυχώς ε, μόνο αφού έχει ε, κλονιστεί η εμπιστοσύνη αρχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα. Πρέπει να δώσουμε ύψιστη σημασία στην ποιότητα και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Φερέρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια συνέβησαν πολλές περιπτώσεις απάτης στην διατροφική αλυσίδα μπροστά στην αποτυχία συστημάτων ελέγχων. Το κρέας το οποίο είχε μολυνθεί με διοξίνες ε, που πέρασε στην τροφική αλυσίδα μέσω προϊόντων ε, ζωικών ε, με τρόπο μη εγκεκριμένο. Και επίσης η νόθευση αλκοολικών προϊόντων, υνοπνευματοδών προϊόντων και όλα αυτά. Είναι σκάνδαλα τα οποία δείχνουν το πόσο παραβιάζονται οι βασικές αρχές της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ποιότητας των τροφίμων απάτες που όχι μόνο αφορούν ελλείψεις ε, του συστήματος ε, ελέγχων αλλά κυρίως ε, συνδέονται άμεσα με την απορρίθμιση και φιλελευθεροποίηση των γεωργικών πολιτικών και εμπορικών πολιτικών με την διεύρυνση αυτών των φαινομένων στη διατροφική αλυσίδα και στις εξαγωγές που ευνοούν τις μεγάλες αγροβιομηχανίες εις βάρος της μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης. Δεν φτάνει μόνο να μιλάμε για ελέγχου. Συνεχίζουν τα σκάνδαλα και αποκαλύπτονται εφόσον αυτά τα πρότυπα δεν αλλάζουν εκ βάθρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερέρα. Δίνω το λόγο στην κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό αφορά την απάτη για τα τρόφιμα και τις διατροφικές κρίσεις. Είναι ένα προφανές ε, θέμα, αλλά οι πιο προφανείς λύσεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Αυτό θα συνιστούσα να κάνουν οι συναδελφοί Ούγγροι. Πηγαίνετε με το καλάτι σας στην αγορά κάθε Σάββατο πρωί και αποφύγετε τις πολυεθνικές που πουλούν ούτως ή σκουπίδια. Υπάρχουν πάρα πολλές αγορές ε, στην Ουγγρική πρωτεύουσα που πολλούν για παράδειγμα ψωμί. Διάφορα προϊόντα τα οποία απολούνται απευθείας από τον παραγωγό. και έτσι αποφεύγουμε το να φτάνουν ε, κακή ποιότητα προϊόντα στο σπίτι μας. Ε, δεν είναι τα προϊόντα αυτά πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ ή από τα διάφορα καταστήματα λιανική. Προσπαθήστε αυτή τη λύση και πάμε όλοι μαζί στην αγορά το Σάββατο. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Πέτροβιτ. The EU has always emphasized the scope. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα επεσήμανε την προστασία των καταναλωτών ως πολιτική προτεραιότητα. Οι πρόσφατες απάτες στον τομέα των τροφίμων διακυβεύουν όχι μόνο την προστασία αλλά και την υγεία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα που βρίσκουν στα αράφια των καταστημάτων ανταποκρίνονται στις δηλώσεις περιεχομένου των προϊόντων αυτών. Έχουν γίνει πολλά ήδη. Έχουν επιτευχθεί πολλά, αλλά παρατηρούμε ότι οι ορισμένοι επιχειρηματίε μπορούν να κάνουν πολλά και διάφορα για να επιτύχουν υψηλά κέρδη. Η πρόσφατη περίπτωση τη εσφαλμένη ε, επισήμανση ε, ζωικών ειδών είναι ε, μια χαρακτηριστική περίπτωση. Παρότι πρόκειται για μεμονωμένε περιπτώσει, Κάθε φορά που αποκαλύπτονται επηρεάζουν πάρα πολύ την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι καταναλωτές οι οποίοι αξίζουν πιο αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς με τελική κατάληξη την πρόληψη παρόμοιων απατών. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ομιλήτρια, κυρία Μπόρζα. svinjsko meso u prodaji kao govedina lano maslinovo ulje pokvareno meso sa svjeim deklaracijama κρέας που πουλείται ω βόηο ή χαλασμένο κρέας που πουλείται ω φρέσκο αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε το 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε αναγκασμένοι διότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία διατροφή δεν ήταν ποτέ χαμηλότερη αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ Στη ΣΥΠΑ, στην Ευ... Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην ΣΥΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συγκεκριμένη περιγραφή τη απάτη των τομέα των τροφίμων. Απλά αναφέρεται κάποιε γενικότητε. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ο ορισμός της απάτης στον τομέα των τροφίμων πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η ποιότητα του ίδιου προϊόντος διαφέρει ανάλογα με το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να έχουμε πολίτε πρώτη και δεύτερη κατηγορία σε μια ενωμένη αγορά. Καλωσορίζω λοιπόν αυτή την έκθεση και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει την κερδοσκοπία ει βάρο τη υγεία μας. Τον λόγο έχει ο επίτροπο ο κ. Ποτόσνικ. Ευχαριστώ τον κύριο Συγητή, τον κύριο Λάγκη και τους συνεισηγητές για τη σκληρή τους δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως την άποψη ότι η αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα αποτελεί για μας προτεραιότητα. Αν θέλουμε βεβαίω να διατηρήσουμε ψηλά επίπεδα ασφαλείας τροφίμων και εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ευρωπαϊκά τρόφιμα και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων. Η Κομισιόν ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες μετά από την αποκάλυψη της απάτης με το κρέας αλόγου πέρσι. Η σχετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της απάτης και στην προσπάθεια πρόληψης και έγκαιρου των απατών στην αλυσίδα τροφίμων. Τόσο τα κρατημέλη όσο και η Κομισιόν συνεργάζονται λοιπόν στον τομέα αυτών, στον εντοπισμό λοιπόν της ε, απάτης και αυτό γίνεται με καλύτερο συντονισμό. Μια ειδική ομάδα δημιουργήθηκε μάλιστα εντό τη ε, γενική διεύθυνση καταναλωτών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντονίσει τι σχετικέ ενέργειε και να συζητά με άλλου αρμόδιους φορείς όπως η Europol τι βέλτιστες μεθόδου για την καταπολέμηση τη απάτη στον τομέα. Επίσης, συζητούμε διάφορες άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης που δρομολογήθηκε πέρσι. Οι τομείς δράσης συνάδουν άλλωστε με την συλλογιστική διέπει τη σημερινή γνωμοδότηση. Προσπαθούμε λοιπόν να εντοπίσουμε μεταξύ άλλων αδήλωτες πόσορτες κρέατος αλόγου σε προϊόντα κρέατος αλλά όπως είπα συζητούμε και άλλες πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την σχετική πρόοδο. Όσον αφορά την προέλευση του κρέατος, προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες νομοθετικής φύσεως για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Μεταξύ αυτών θα συμπληρωθεί το σύνολο υποχρεώσεων επισήμανσης για το χείρινο κρέας, το βόλιο και το κρέας των πουλερικών. Το ίδιο ισχύει και για τις, περιπτώσεις όπου το κρέας χρησιμοποιείται ως συστατικό άλλων τροφίμων. Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορεί να ικανοποιούν την ανάγκη εντοπισμού της πρόληψης, την ανάγκη ίχνη όμως τα μέτρα αυτά δεν θα εξαφανίσουν την απάτη. Το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου μας δείχνει ότι ακόμη και αν η υποχρέωση επισήμανση ίσχυε είναι εκείνη την εποχή, δεν θα είχαμε αποφύγει την απάτη. Όσον αφορά την κλωνοποίηση, στι 18 Δεκεμβρίου η Κομισιόν υιοθέτησε δύο προτάσει. Η μία αφορά την προστασία των ζώων σχετικά με τις τεχνικές κλωνοποίησει. Με την άλλη πρόταση απαγορεύεται η κλωνοποίηση των εκτροφωμένων ζώων και απαγορεύονται οι σχετικέ αγωγέ. Απαγορεύονται επίση το κρέα και το γάλα από τέτοια ζώα και απαγορεύεται η διαθεσή του στην κοινωτική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει ο πρόεδρο. Πέρα τη συζήτηση, η ψηφορία αύριο στι 12. Και τώρα προχωρούμε. Έκθεση Steinruck αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Δίνω τον λόγο